Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρωτού ε, before ε, να καλωσορίσω και να δώσω το λόγο στους αξιότιμους ε, προσκεκλημένους να πω ότι υπήρξε μία συμφωνία μεταξύ των μελών. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το σημείο 16 διότι ο εισηγητής ο κύριος Καβαντά θέλει να φύγει νωρίς γιατί έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Αν δεν υπάρχει λοιπόν αντίρρηση δίνω το λόγο κατευθείαν στον κύριο Καβαντά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση σχετικά με αυτό που ήδη είχαμε συμφωνήσει στα τέλη του σήμερα. Σας είχα πει, τέλη, στο τέλη του πρωινού σας είχα πει ότι είναι ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Οι ακροάσεις ε, στην αρχή της νομοθετικής περίοδου όπως θυμάστε έγιναν πέρυσι το καλοκαίρι και μας κατέστησαν δυνατό να διαπιστώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη θέση που περιμένει ε, ο κόσμος να έχουμε. Και συγκεκριμένα εμείς προσπαθούμε να δούμε τις, ε, τους καλύτερους τρόπους για να νομοθετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση γενικά θέλουμε ε, με κάποια εργαλεία που έχουμε να βλέπουμε πόσο ειλικρινής είναι η Επίτροπη στις δηλώσεις τους. Ας πούμε σε δύο-τρεις περιπτώσεις που είχαμε πολιτικά ζητήματα αλλά υπήρχε και μία περίπτωση που είχαμε θέματα τεχνικά, ειλικρίνειας δηλαδή. Όμως ε, η διαδικασία δεν είναι αρκετά διεξοδική και μπαίνουμε σε μια ζώνη αβεβαιότητας. Δεν ξέρουμε τι βρίσκεται πίσω από μια δήλωση αν εγώ ήμουν υποψήφιος ας πούμε ε, επίτροπος και ήθελα να ασχοληθώ με την αυτοκινητοβιομηχανία ας πούμε και ήθελα να πάρω το χαρτοφυλάκιο της αυτοκινητοβιομηχανίας και ε, των μεταφορών. Αν είχα κάποια συμφέροντα οικονομικά θα τα πούλαγα, αλλά θα τα πούλαγα στην αδελφή μου, τη μάνα μου, την ε, γυναίκα μου, ε, εγώ βέβαια δεν έχω οικογένεια, εγώ είμαι οικογένεια, αλλά εντάξει. Γενικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ε, γιατί δεν μπορούμε να δούμε ακριβείς και συγκεκριμένες πληροφορίες για την ειλικρίνεια και για τη βάση επί της οποίας γίνονται αυτές οι δηλώσεις. Ε, και εμείς ως βουλευτές όταν βάζουμε την υπογραφή μας δεν πρέπει να είμαστε παγιδευμένοι από ψέματα τα οποία γίνονται από παράληψη βέβαια. Για παράδειγμα, υπήρξε κάποιος επίτροπος ο οποίος όντως δήλωσε ε, για τα οικονομικά του συμφέροντα ότι τα είχε πουλήσει, αλλά δεν είχε δηλώσει σε ποιον τα είχε πουλήσει. Οπότε υπήρξε μια συγκεκριμένη διασταύρωση των οικονομικών συμφερόντων λοιπόν. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα πρέπει να διατηρήσει τις αρμοδιότητές της για την εξέταση των οικονομικών συμφερόντων αλλά θα πρέπει να έχει και πραγματική εξουσία είτε η ίδια αλλά αυτό είναι μάλλον λίγο πολύπλοκο ή να δώσει την εντολή σε κάποιον ε, ικανό ε, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες οργανώσεις που μπορούν να διερευνήσουν και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ας πούμε επιμελητήριο σχετικό το οποίο να βρίσκεται ας πούμε στην Όλαφ ε, που ασχολείται με την πάταξη της απάτης και να μπορεί να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, όπως για παράδειγμα μας είπε ο κύριος Ναντάλ, υπάρχουν πολλά τέτοιοι θεσμοί στην Ευρώπη. Μπορούμε λοιπόν να ε, μάθουμε από τα μαθήματα του 2014 με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων για να μπορεί η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων όχι να έχει περισσότερες εξουσίες εναντί των άλλων, αλλά να έχουν πραγματικές εξουσίες, ε, να τιμάται η υπογραφή της και να γίνεται, σεβαστή, γίνεται σεβαστός ο ρόλος τους. Δεν είναι ότι δεν γίνεται σεβαστός ή ότι δεν είμαστε ειλικρινείς ή δεν έχουμε το θάρρος, αλλά δεν έχουμε τα εργαλεία τα κατάλληλα για να πάμε σε βάθος αυτές τις έρευνες. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό είναι ένα θέμα και μπορούμε να έχουμε και ένα σεμινάριο με τη μορφή που θέλετε και να σκεφτούμε έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο των ε, ε, επιτρόπων να είναι αντίστοιχα με αυτά των βουλευτών. Ποια είναι η δημοκρατία που λειτουργεί σωστά. είναι μια εκτελεστική εξουσία ε, η οποία έχει αντίστοιχα και νομοθετικές επιτροπές οι οποίες ε, μπορούν να κρίνουν ε, τεχνικά για, επί των θεμάτων και να ψηφίζει και πολιτικά βέβαια. Αυτό είναι μια ολοκληρωμένη δημοκρατία. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο σεμινάριο με συνταγματολόγους, Ευρωπαίους που έχουν μια μεγάλη παράδοση δημοκρατική εδώ 15, 20, 25 χρόνια και οι φίλοι μας οι Πολωνοί είναι πραγματικά ένα ε, εξαίρετο παράδειγμα στον κόσμο από μια τυραννία που πηγαίνουν τώρα ε, που πήγαν τόσο γρήγορα σε μια δημοκρατία. Είχαμε ας πούμε περιπτώσεις ε, γκάγκστερ το 70 με τον κύριο Μούγκα, αλλά αυτό ήταν συγκεκριμένο επεισόδιο. Τέλος πάντων είναι τώρα όμως αρκετά όριμοι στην Ευρώπη για να μπορούν να προσπαθούν τα χαρτοφυλάκια των επιτρόπων να συμπίπτουν με αυτά των επιτροπών ε, του Κοινοβουλίου για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, ε, το να πρέπει μία επιτροπή να ασχολείται με ένα πρόβλημα μέσω διαφόρων ε, επιτρόπων. Το είχαμε δει αυτό στην προηγούμενη νομοθετική περίοδο και αυτό ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο γιατί υπήρχε το συνδικάτο του του τρόμου. Πρέπει να σταματήσει αυτό, πρέπει πραγματικά τα χαρτοφυλάκια των ε, επιτροπών να συνάδουμε αυτά των επιτρόπων ή το αντίθετο έτσι ώστε να υπάρχει πραγματικός έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας. Ε, εδώ λοιπόν ε, ολοκληρώνω για αυτό το σεμινάριο ή έστω μια ακρόαση τριών-τεσσάρων ωρών με συνταγματολόγους για να μπορεί να προταθεί στο Κοινοβούλιο ε, ποια είναι σωστή διαδικασία. Ξέρουμε ότι η βασική μας εχθρή είναι η αποχή και η ακραίοι, αλλά η ακραίοι δεν είναι ε, κατά τύχη ακραίοι ε, και δεν πρέπει όλους να τους κατηγορούμε γιατί ανταποκρίνονται σε ανάγκες των εκλογέων. Άρα είναι ένα τεράστιο θέμα που θα πρέπει να το ανοίξουμε ε, γι' αυτό σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι που ε, δεχτήκατε να με ακούσετε. Ο κύριος Ζήσκα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. ευχαριστώ Σαμάρη Καβαντά. Ευχαριστώ συνάδελφε για την ορθή παρουσίαση αυτού του σημαντικότατου θέματος. Θυμόμαστε ακόμη το ακαθόδες μονοπάτι που έπρεπε να διανύσουμε κατά τη διάρκεια των ακροάσεων και θα χρειαστεί μία περίοδος περισυλλογής. Έχουμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε για νέα δράση για το 2019 όταν θα υπάρχει το νέο σώμα των επιτρόπων και θα πρέπει να γίνει και από τα τρία θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και το Συμβούλιο. <coughs> Φυσικά το πιο ενδιαφέρον είναι οι δικέ μα αρμοδιότητε και το δικό μα συμφέρον, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να συμμετέχουμε σε αυτέ τι ακροάσει και θα πρέπει επίση να εγκρίνουμε ε, την οποιαδήποτε <clears throat> διάταξη της ε, εκάστοτε επιτροπής. Χρειαζόμαστε πιο λεπτομερείς αλλά και πιο σαφείς σχέσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και ε, την Επιτροπή τις επιτροπές ανάλογα με τις αρμοδιότητες των εκάστοτε επιτρόπων. Γνωρίζετε, το έχω επαναλάβει πολλές φορές, ότι δεν θέλω αυτή μας η επιτροπή να γίνει ένα διερευνητικό όργανο, όργανο διερεύνησης, ανακριτικό. Αλλά, Ζαμαρή, συμφωνώ μαζί σου και έχει αναφερθεί και στην Όλαφ. Ίσως η Όλαφ, ε, το γραφείο τη απάτης, θα μπορούσε να ελέγξει τις ε, τοποθενέσχες ε, των μελλοντικών επιτρόπων και θα μπορούσα και εγώ να ε, προγράψω αυτό. Θα πρέπει να θυμόμαστε βέβαια ότι τώρα πρέπει να αναπτύξουμε κάποια διαδικασία για τις ακροάσεις των επιτρόπων. Αλλά αυτό έχει σχέση και με άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, την διάταξη, την σύνθεση αυτής της Επιτροπής, της Κομισιόν. Αγαπητοί φίλοι, λοιπόν, ε, είμαι Είμαι υπέρ της συνθήκης, της συνταγματικής συνθήκης και δούλεψα πολύ σκληρά στην Πολωνία για να προωθήσω αυτή την ιδέα και η Πολωνία θα είχε αποδεχτεί αυτή την συνθήκη. Δυστυχώς όμως οι Γάλλοι φίλοι μας απέρριψαν ε, στο δημοψήφισμα αυτή την συνθήκη, θα ήταν οι πρώτοι και μετά ακολούθησαν και οι Ολλανδοί. Και αυτό είναι απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά είναι αλήθεια ότι σε ένα κολέγιο 28 ανθρώπων, ε, που ίσως να είναι ακόμα μεγαλύτερο στο μέλλον, αν δεν αλλάξει τίποτα είναι παράλογο. Κάποιες φορές δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Κάποιες φορές ε, μπορεί να χρειάζεται κανείς να λάβει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και η προσπάθεια από την Επιτροπή Γιούγκερ δεν μπορεί πραγματικά να αξιολογηθεί αυτή τη στιγμή διότι είναι ένα σημείο έναρξης απλώς οπότε δεν, δεν γνωρίζουμε ακόμα τον καταμερισμό των εργασιών. Υποτίθεται ότι είχαν μείωση του αριθμού των χαρτοφυλακίων και των επιτρόπων αλλά υπάρχει πολλή δρόμος ακόμα γι' αυτό. Αν κοιτάμε λοιπόν ε, τις καθημερινές εργασίες του Κοινοβουλίου, αν δούμε λίγο και την ακρόαση που προτείνατε, το να είναι η Κομισιόν ε, συνδεδεμένη με μια αντίστοιχη, ένα, ένας, κάθε επιτροπή συνδεδεμένη με έναν μόνο επίτροπο, ε, τότε δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό, γιατί πολλές φορές το πεδίο είναι πάρα πολύ ευρύ για τα, στα διάφορα ζητήματα. Οπότε μπορεί να χρειάζονται τρεις-τέσσερις επιτροπές. Οι ακρόασει θα πρέπει να γίνονται σωστά, σίγουρα, αλλά ε, δεν μπορούμε να κάνουμε έναν εξορθολογισμό όπως θα θέλαμε, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπαρχουν τρει τρει-τέσσερι επιτροπές που να θέλουν να ακούσουν έναν υποψήφιο επίτροπο. Στην ουσία λοιπόν δεν θα έπρεπε να έχουμε αυτή τη διασπορά των καθηκόντων. Ξέρουμε ότι όταν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν τρεις διαφορετικές επιτροπές, έχουμε και τρεις διαφορετικές γνώμες γνωμοδοτήσεις. Οπότε, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για τα τρία θεσμικά μας όργανα και να δούμε πώς μπορούμε να προλαμβάνουμε τα πιθανά προβλήματα. Χαίρομαι που ξεκινάει τώρα αυτή η δουλειά γιατί θα έχουμε αρκετό χρόνο για να συνεχιστεί η ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε ένα τελικό προϊόν εκ μέρους του ΕΛΚ και ως σκιώδης εισηγητής θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Καβαντά Ε, ήμουν εδώ σε δύο ακροάσει, ε, στην πρώτη συγκεκριμένα, είδα πραγματικά ότι θα μπορούσαν οι ευρωβουλευτές να έχουν έναν πραγματικό ρόλο, αλλά αυτός ο ρόλος πρέπει πραγματικά να αναθεωρηθεί. Και ο κύριος Καβαντά το έθεσε σωστά το ζήτημα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ίδια τη διαδικασία. Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι επίτροποι κάνουν μια παρουσίαση και μετά εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις. Όμως όλα αυτά ε, είναι πολύ τυποποιημένα, άρα δεν υπάρχει πραγματική δυνατότητα ε, για να θέσουμε ουσιαστικές ερωτήσεις, αλλά γιατί όλα είναι προετοιμασμένα από πριν και δεν μπορούμε να φτάσουμε στα πραγματικά ζητήματα. Και όπως γνωρίζουμε δεν είναι και τόσο δύσκολο αν βάλεις χρόνο και προσπάθεια ε, μπορείς να προετοιμάσεις αυτό που θες να απαντήσεις και έτσι δεν μπορούμε να, δούμε τι θέλει και τι δεν θέλει να κάνει ο Επίτροπος. Η οργάνωση είναι δύσκολη γιατί και για τους ευρωβουλευτές είναι δύσκολο αλλά θα ήθελα να έχουμε χρόνο για ερωτήσεις και για συμπληρωματικές ερωτήσεις επιπρόσθετες για να δούμε ποια είναι η πραγματική γνώμη των επιτρόπων για τα διάφορα ζητήματα. Κομμάτι αυτού και είναι κάτι που δεν συζητείται τόσο πολύ ε, είναι νομίζω η διαδικασία με την οποία ψηφίζουμε όλη την Επιτροπή. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ρεαλιστική άποψη και να αναλαμβάνει κανείς ε, δράση γιατί πρέπει να στραφείς εναντίον όλων. Και στην τελευταία εντολή υπήρχαν πάντοτε τρόποι για να το παρακάμψουμε αυτό, Α πούμε το κράτος μέλος έβρισκε κάποιον άλλον να αντικατασταθούν οι προβληματικές περιπτώσεις, αλλά δεν είναι αυτό ικανοποιητικό. Ίσως καλό θα ήταν να είχαμε και στην Ολομέλεια τη δυνατότητα να ψηφίζουμε ξεχωριστά για κάθε επίτροπο και όχι για όλο το κολέγιο. Επίσης θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα του αριθμού των επιτρόπων, ανάλογα με την καταγωγή τους. Ας πούμε, είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν δύο-τρία κράτη-μέλη για να προτείνουν ένα συγκεκριμένο, έναν και μόνο επίτροπο. Βέβαια, 28 επίτροποι είναι πάρα πολλοί ε, και όπως είπε ο κύριος Ζήφκα, έτσι φτιάχνουμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, μόνο και μόνο για να έχουν κάτι να κάνουν. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους ε, και γενικά η μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ των ε, χαρτοφυλακίων των Επιτρόπων και των Επιτροπών του Κοινοβουλίου θα ήταν καλό, γιατί είναι δύσκολο. Αυτό που κάνει η Επιτροπή ε, αλλάζει σε κάθε εντολή. Είναι διαφορετικό αυτό που κάνει η Επιτροπή Γιούνκερ από την Επιτροπή Μπαρόζο. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και να σεβόμαστε το ίδιο το κοινοβούλιο και τον τρόπο σύστασης των επιτροπών, γιατί δεν θέλουμε στην ουσία να έχουμε χαρτοφυλάκια και ευθύνε και αρμοδιότητες που να αλλάζουν και για τις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Χρειάζεται πολύ σκέψη λοιπόν γι' αυτό. Και τέλος, όλα αυτά για τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων και το ρόλο αυτής της Επιτροπής κατά την εξέταση αυτών των δηλώσεων. Στην αρχή αυτής της ε, θητείας υπήρχαν ε, πάρα πολλά ζητήματα που τέθησαν για ένα συγκεκριμένο επίτροπο και κάποιοι από εμά θεώρησαν ότι αυτή η επιτροπή θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να θέτει περισσότερες ερωτήσεις για να ανακαλύπτει περισσότερα στοιχεία. Αυτό δεν είναι κριτική, απλώς θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει λίγο παραπέρα σε αυτή την Επιτροπή για, αυτό το, για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση από ό,τι πήγαμε. Το να μιλάμε για να ανακριτικές εξουσίες ε, είναι βαρύ στα αγγλικά τουλάχιστον. Δεν ξέρω στις άλλες γλώσσες λέει ο Μιλήτρη. Γενικά θα είναι καλό να έχουμε δυνατότητα εξέτασης και γενικά να είναι λίγο παραπάνω υπέρ οι δυνατότητε μα από ό,τι έχουμε τώρα. Αλλά σα ευχαριστώ κύριε Καβαντά και τον κύριο Κόρπετ για μια πολύ χρήσιμη έκθεση κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκούτλαντ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να στηρίξω του ε, συναδέλφου στην Επιτροπή. Νομίζω έχετε αφήξει εξαιρετικά τα σημεία για το ποιο θα μπορούσε να ήταν ο ρόλο μα και πώ θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε. Πιστεύω το θέμα του το πώς να γίνονται πιο σαφείς οι δηλώσεις όταν έχουμε ένα πρόβλημα με έναν επίτροπο, θα πρέπει να είναι ευκολότερο αν βρούμε έναν τρόπο να ψηφίζουμε διαφορετικά προτού ψηφίσουμε για ολόκληρο το σώμα των επιτρόπων. Νομίζω αυτή είναι πολύ καλή ιδέα. Επίσης θα ήθελα και εγώ να προσθέσω ένα πρόβλημα σχετικά με την ισότητα γυναικών ανδρών. Επειδή ε, τα κράτη-μέλη δεν διορίζουν με ισότιμο τρόπο, έχουμε πρόβλημα να έχουμε ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα στην Επιτροπή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα, να το κάνουμε πιο ισορροπημένο. Ίσως θα πρέπει να αναζητήσουμε ε, τρόπους έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να ορίζουν δύο άτομα και είναι σημαντικό να λεχθεί ως ε, ρόλος μου ως εισηγήτρια για τα θέματα φύλων και ισότητας ε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό να συζητηθεί. Ο κ. Ντυρό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εντάχει να πω βέβαια ότι το θέμα των, του, των δύο φύλων είναι ένα, πραγματικά ένα ζήτημα το αν πρέπει να έχουμε ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες ε, στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο είναι επίσης ε, ζήτημα. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι στην Κομισιόν υπάρχει ένας εγκάρσιος χαρακτήρας που δεν αντανακλάται ε, σε εμά. Θα πρέπει να το σκεφτούμε. Θα, θα, ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καβαντά για την, το αξιοθαύμαστο έργο του. Αυτό το έγγραφο είναι, θα έλεγα, 100% ε, ε, εξαιρετικό. Δύο παρατηρήσεις μικρές ε, σε σχέση με αυτό που έγινε στις αρχές των ακροάσεων. Πρώτον, θα επιθυμούσα να μπορούσαμε να σκεφτούμε την εναρμόνιση της δήλωσης ενδιαφέροντος με τη χάρτα καλής συμπεριφοράς γιατί εκεί ε, υπάρχει μια αναντιστοιχία και θα μπορούσε να δει, θα πρέπει να διευκρινιστεί ή θα το αφαιρέσουμε ή θα το βάλουμε παντού, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει σε μία, στο ένα γράφο και να μην υπάρχει στο άλλο. Θα υπάρχει, πρέπει να υπάρξει κάποια αναρμόνιση. Το δεύτερο ε, για, ε, για την υπεράσπιση της Κομισιόν μας έγιναν αρκετές ε, συζητήσεις για το θέμα του σκρούτινη, του, της εξέτασης, του ελέγχου. Ε, υπάρχει μια ισχυρή βούληση όπως το Κοινοβούλιο να, να παίξει το ρόλο του στο τέλος της ε, έρευνας της εξέτασης ε, θα ήθελα να, μην η, Κομισιόν να μπορεί να βλέπει και τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. Άρα η εξέταση από την αρμόδια επιτροπή και η ακρόαση του επιτρόπου μπορεί να γίνεται μόνο αφού ε, του ε, ξεκαθαρίσει το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. του γίνει ακρόαση του Επιτρόπου. Είναι κάτι το οποίο επίσης εκφράσαμε και την τελευταία φορά. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Καβαντά, θέλετε να συνοψίσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Βλέπω ότι μετά την ε, πρώτη φάση που είχαμε το 2014 που ήμασταν κάπως στριμωγμένοι ε, με θέματα που, όπου νιώθαμε ότι δεν ήμασταν επαρκείς και δεν είχαμε ε, τη δυνατότητα να τα αναλάβουμε. Πραγματικά τώρα σας ευχαριστώ που όχι μόνο εμπλουτίσατε αλλά έχετε ουσιαστικά κτίσει πάνω ε, στην ταπεινή μου πρόταση. Θα ήθελα, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω σε συντομία στους τρεις συναδέλφους, τέσσερις συναδέλφους που παρενέβησαν, ε, τον κύριο Ζήσκα που θα ήθελα να ευχαριστήσω, θα ήθελα να πω ότι έχει δίκιο. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την οδό της μίας εκτελεστικής ευθύνης που να ελέγχεται από την νομοθετική αρμοδιότητα. Όλες οι χώρες που λειτουργούν καλά δημοκρατικά είναι έτσι φτιαγμένες. Και ξέρετε ότι σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου, τις πραγματικές, η Επιτροπή Νομική είναι το άτομο, το, το, το κέντρο των πολιτικών συζητήσεων και μπορούμε να γίνουμε με την βάθυνση των, ε, του θεσμού της λειτουργίας μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Μονεπόλ, την άκουσα με πολύ ενδιαφέρον γιατί ε, ένα Κοινοβούλιο έχει πολύ σημαντικές ευθύνες στην πλάτη του. Αλλά όταν γνωρίζουμε τις εργασίες της εσωτερικές, ξέρουμε ότι πολλές φορές ε, κοιτάμε ε, επιφανειακά ορισμένα πράγματα ή ε, άλλους συναδέλφους ή όμως υπάρχουν κάποιες ζώνες πολύ σημαντικές που ε, μπορούν να ε, δώσουν μια αρνητική εικόνα στην φήμη μας. Για να μιλήσουμε τώρα σαφώς, όταν υπάρχουν προβλήματα συγκρούσεων, σοβαρών συγκρούσεων και θέματα που συζητήσαμε σήμερα, άρση ε, της ασυλίας του τάδε ή του δίνα. Έχουμε ε, όταν έχουμε συμφέροντα μιας ε, γνώμης κατά μιας άλλης. Θα πρέπει να ξέρουμε αν έχει υπάρξει απάτη, αν υπάρχει πλουτισμός, αν υπάρχει ψέμα ε, ή αδίκημα. Ε, μια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων σε όλα τα κοινοβούλια και είναι, έχει ανάγκη να έχει ένα φορέα έρευνας εμείς είμαστε ένας μεγάλος μηχανισμός, αλλά θα πρέπει να είναι στην διάθεσή μας ε, και να αναθέτουμε ε, την εξέταση διαφορών θεμάτων. Γι' αυτό έχω σκεφτεί την Όλαφ που υπάρχει, αλλά όπου ε, πρέπει να προσθεθεί ένας, μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Και αυτό θα αυξήσει την αξιοπιστία του ρόλου μας αν στο τέλος αυτής της θητείας θα μπορούμε να δείξουμε ότι είμαστε πολιτικοί κριτές αλλά δίκαιοι κριτές σε πολιτικά θέματα και εμπνέουμε τους ε, ψηφοφόρους μας. Αλλά ε, ότι στηριζόμαστε σε ένα όργανο έρευνας που είναι αδιαμφισβήτητο ανεξαρτήτως ε, πολιτικού χρώματος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το θέμα κυρία Μάνιπολ. Το Κογκρέσο, το Αμερικανικό και μιλάω τώρα για τη μορφή του, το ξέρετε περισσότερο. Εγώ ε, δούλεψα όταν ήμουνα και δημοσιογράφος στην Washington, το Κογκρέσο έχει μια πολύ απλή μέθοδο λειτουργίας. Όταν κάποιος εμφανίζεται ενώπιό τους, εάν δεν έχουν εξαντλήσει όλα τα θέματα, το άτομο το οποίο εμφανίζεται ενώπιό τους, είναι στη διάθεση να δώσει απαντήσεις. Δεν είναι 20 λεπτά. Αν χρειάζεται μια μέρα, θα πάρει μια μέρα. Και νομίζω θα πρέπει να το ακολουθήσουμε. Και για να κλείσω θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντυρό για αυτά που είπε. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω, γιατί και εσείς και εσείς κυρία ε, πραγματικά ε, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την ε, πρότασή μου και ε, τέλος είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα θα πρέπει να κάνουμε μόνιμο σεμινάριο μέχρι το τέλος αυτής της θητείας ένα άτυπο σεμινάριο που ε, από καιρό σε καιρό θα καλεί ε, αυτούς ε, που ε, είναι στη διάθεσή μας να είναι άτυπης μορφής και στο τέλος της θητείας θα έχουμε μια δεύτερη έκθεση έτσι ώστε να μπορούμε να νομοθετήσουμε σε εισαγωγικά και να μπορούμε να εξετάσουμε όλα αυτά που θα κάνουν τον θεσμό μας να προοδεύσει. Δεν ξέρω αν δέχεστε αυτή την ιδέα. Δεν περιορίζει κανέναν, αλλά θα έχουμε την πολιτική ευχαίρεια να αποφασίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Καβαδά. Και τώρα θα περάσω στην Αγγλική. Ευχαριστώ κύριε Καβαδά. Τώρα επανερχόμαστε στο σημείο 13 της Συνδυσίας Διάταξης Έχω την τιμή για μια ακόμη φορά να καλωσορίσω εκπροσώπους του ELI, Ευρωπαϊκού του Δικαίου και θα μας κάνει μια παρουσίαση σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες πολιτικής δικονομίας. Ε, Παραβρίσκεται επίσης και το UNIDROIT Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου και συναδέλφους από το UNIDROIT για να σας εξηγήσουμε ομού το σχέδιο που θέλουμε να προωθήσουμε σχετικά με τους κανόνες της πολιτικής δικονομίας. Γνωρίζω πως ε, ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο, η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες στην Ένωση πρόσβαση σε αυτήν αλλά και στις επιχειρήσεις. Ε, κανείς καλύτερα από τα μέλη της Επιτροπής σας δεν γνωρίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν στις διάφορες εθνικές νομοθεσίες και εθνικές κουλτούρες προκειμένου να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο πρόσβασης στην δικαιοσύνη. Του του λεχθέντος φυσικά υπάρχουν μια σειρά από νομικά εργαλεία που αφορούν την πολιτική δικονομία όπως ε, η όπως το θέμα των διαδικασία μικροδιαφορών, διαδικασία της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως κάποιες οργανώσεις που στο παρελθόν παρατήρησαν ότι το ε, Ινστιτούτο Αμερικανικής Νομοθεσίας μαζί με την UNIDROIT το 2004 κατόρθωσαν να καταρτήσουν αυτό το έντυπο που αφορά στις εθνικές νομοθεσίες. Πρόκειται για soft law, ενδοτικό δίκαιο και αφορά στη, στην νομοθεσία και στα δικαστήρια, τα εθνικά δικαστήρια. Θεωρήσαμε όμως ότι θα ήταν ορθό και επίκαιρο να προβούμε σε μια παρόμοια σε ένα παρόμοιο εγχείρημα και στην Ευρώπη Λοιπόν, λαμβάνεις υπόψη αυτά ως έμπνευση. Συστήσαμε μια σειρά από ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, νομικοί, δικαστικοί, προκειμένου να παράγουμε νομοθεσία στο ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκή Ένωση και να απλουστεύσουν τις ε, διαδικασίες ε, πολιτικής δικονομίας. Ε, εδώ και 18 μήνες δουλεύουμε πάνω στο ζήτημα. Οι συνάδελφοι μας στην Κομισιόν έδειξαν ενδιαφέρον για τις εργασίες και τις παρακολουθούν εκ του και ακούσαμε με ικανοποίηση ότι και εσείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα αναλάβετε μια πρωτοβουλία από την κατεύθυνση αυτή. Τώρα αυτά περί εισαγωγή. Έχω εδώ τρεις από τους εισηγητές σήμερα, οι οποίοι η συντομία θα σας εξηγήσουν το θέμα της ε, παράδοση εγγράφων και ο συνάδελφός μου από το Unit θα προσθέσει κάποια λόγια. Αυτά και ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε στην σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ, με ακούτε. Θα σας μιλήσω για την επίδοση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, είναι τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον της Επιτροπής σας για να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση του σχεδίου ε, με το οποίο ασχολούμαστε. Είμαι μία από τις συνεισηγήτριες της ομάδας που ασχολείται ή προσπαθεί τέλος πάντων να θεσπίσει κανόνες για την επίδοση των εγγράφων ε, και την ενημέρωση για την έναρξη δικαστική διαδικασίας. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που σχετίζονται με αυτά που είπε η Νταϊάννα. Φυσικά από την αρχή αυτού του project ε, συζητήσαμε πάρα πολύ το εύρος, το πεδίο και για να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινεί εξ αυτό το πεδίο είναι ρευστό. Διότι είμαστε μια ανεξάρτητη ομάδα ανθρώπων και δεν έχουμε εξ αρχής ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, αλλά η κάθε ομάδα όπως εργάζεται βρίσκει ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το πεδίο της και το συζητάμε και το θεσπίζουμε αντίστοιχα. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε κάποια μορφή βέλτιστων πρακτικών στην ε, πολιτική δικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να χτίσουμε πάνω σε αυτά που έχει ήδη κάνει το ELI και το UNITROA. Επειδή είναι πρότυπο νομοθεσίας, ε, έγιναν πολλές συζητήσεις στις ομάδες ε, που ασχολούνται με το θέμα αυτό και συζητήσαμε για το πώς πρέπει όλα αυτά να σχετίζονται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ε, συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Βλέπουμε ότι ο ρόλος μας δεν ε, δεσμεύεται υπό μια έννοια από το κεκτημένο, αλλά από τις βέλτιστες πρακτικές για το μέλλον. Φυσικά το κεκτημένο το λαμβάνουμε υπόψη μας και το βλέπουμε ως ε, μια πολύ σημαντική πηγή, αλλά δεν είναι και η μονοδική πηγή έμπνευσης για το project μας. Σε ευρωπαϊκό βέβαια πλαίσιο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε πλήρως. Άλλες πηγές είναι οι κρατικές ε, διαδικασίες πολιτικής οικονομίας ε, και άλλα project ερευνητικά που μπορούν να μας εμπνεύσουν και να συμβάλλουν περαιτέρω στο έργο μας. Ήδη το συζητήσαμε σήμερα κατά τη συνάντηση των ομάδων μας, ποιες πρέπει να είναι οι προοπτικές μας. Είχαμε πολλές συζητήσεις σχετικά με το γεγονός ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε σύγχρονες φυσιολογικές εξελίξεις και να βασιστούμε στις εξελίξεις που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη, τα οποία είναι πιο προηγμένα σε θέματα όπως ας πούμε η τεχνολογία τα συστήματά τους. Αυτό για την ομάδα της επίδοσης ε, είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο. Συγκεκριμένα ε, μιλάω για την ηλεκτρονική επίδοση που πρακτικά και ουσιαστικά είναι ένα σημαντικό ε, θέμα για το μέλλον. Οπότε, Αυτά λίγο πολύ είχα να πω για τις προοπτικές και το πεδίο της ομάδας μας. Ε, ακόμα δεν έχουμε επίσης ε, θεσπίσει το επίπεδο λεπτομέρειας. Όταν έχουμε έναν πρότυπο κώδικα, δεν ξέρουμε αν θέλουμε να περιλάβουμε κανόνες οι οποίοι θέλουν να εμπνεύσουν εσωτερικούς ή διακρατικούς κανόνες. Τώρα επίση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλο ζήτημα το τι είναι κρατικό και το τι είναι διακρατικό. Γενικά, ίσως ε, το σχέδιό μας ε, θα πρέπει να έχει στοιχεία από όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ σε αυτή τη διάκριση. Τα μοντέλα πρέπει να μας εμπνέουν το ίδιο και σε κρατικό και σε διακρατικό επίπεδο. Αν, δεν, αν μπούμε πολύ σε λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα, μπορεί να μην βλέπουμε την ουσία του έργου. Τώρα, όσον αφορά στην επίδοση, γνωρίζω ότι είστε πολύ απασχολημένοι και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό δεν θα μπω και σε υπερβολικές λεπτομέρειες. Αλλά, αν με επιτρέπετε, ήθελα να σας διαβάσω κάτι, γιατί στην ουσία Υπάρχει ένα εναρκτήριο λάκτισμα, αυτό που βλέπετε εδώ. Οι περισσότερες ομάδες από εκεί ξεκίνησαν. Ε, το πολύ ενδιαφέρον ήταν ε, ότι συνειδητοποίησαμε πως αυτούς τους κανόνες ε, που είναι πολύ γενικοί μπορούμε να τους αναπτύξουμε περαιτέρω με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Να σας διαβάσω λίγο όμως κάτι για να πάρετε μια γεύση για το ποια είναι η βασική μας έμπνευση. δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αν το θυμάστε. Στο 5.1, σε αυτό που ονομάζεται αρχές βασικά και όχι κανόνες, λέει στην αρχή της ε, διαδικασίας η ενημέρωση που δίνεται με μέλη τα οποία ε, είναι ευλόγως αποτελεσματικά ε, δεν θα, πρέπει να θα πρέπει να δίνεται σε... με άλλους εκτός του κατηγορούμενου. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς, τις πληροφορίες για τις μεθόδους προσφυγής και τα μέτρα που... και ε, θα πρέπει τα μέρη να ενημερώνονται για τη διαδικασία, για την αντίδραση, την απάντηση που μπορεί να έχουν και ποια θα είναι η επίπτωση αν δεν απαντήσουν εγκαίρως. Και τέλος, τα έγγραφα θα πρέπει να είναι στη γλώσσα του δικαστηρίου αλλά και των ε, ατόμων που έχουν, ε, και, στη, και στη γλώσσα της χώρας όπου τα άτομα έχουν ε, την κατοικία τους ή την ε, επιχειρηματική τους έδρα. Αυτή είναι λοιπόν η αφετηρία για εμάς. Όπως βλέπετε αυτές οι σύντομες αρχές δεν περιλαμβάνονται σε ένα κώδικα πολιτικής δικονομίας για την επίδραση, δίνουν μια γενικότερη κατεύθυνση. Εν μέρει λοιπόν, βάσει αυτού του βιβλίου μπορούμε να δούμε ποια είναι η μορφή πληροφοριών που πρέπει να δίνεται, ποια είναι η μορφή των εγγράφων ε, που θα επιδίδονται, ποια είναι η γλώσσα. Επίσης προσπαθούμε αν μπορούμε να δώσουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες, να εξετάσουμε τις μεθόδους επίδοσης και να δώσουμε κάποια ένδειξη σχετικά με το ποιες μέθοδοι μπορεί να είναι η βέλτιστη πρακτική. Τέλος, να θέσω πάλι ε, ένα θέμα που έχει να κάνει με την ηλεκτρονική επίδοση και τις μεθόδους. Έχουμε εξετάσει πάρα πολύ το πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ηλεκτρονική επίδοση και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε όσο πιο γενικοί γίνεται για να μην δεσμευτούμε ε, από κάποια συγκεκριμένα τεχνολογικά πρότυπα. Η ομάδα μας έχει επικεντρωθεί στο εξή. Όταν χρησιμοποιείς ηλεκτρονικά μέσα, πώς μπορείς να διασφαλίσεις ότι ο κατηγορούμενος θα λάβει τελικά το έγγραφο και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε να γίνει σωστά η επίδοση. Πρέπει να υπάρχει ας πούμε επίσημη συνένεση για να μπορούν να λαμβάνουν τα μέρη ηλεκτρονικά, τα έγγραφα. Γιατί πολλές φορές ε, χρειάζεται τέτοια επίσημη αποδοχή πριν κανείς ε, μπορέσει να επιδώσει ηλεκτρονικά ένα έγγραφο και επίσης πώς θα απαντά κανείς σε μια τέτοια ηλεκτρονική ενημέρωση ή επίδοση με email για παράδειγμα ας πούμε αν κάποιος είναι διακοπές τι σημαίνει αυτό τι εγγυήσει έχουμε ή τι εγγυήσει θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε σε επίπεδο ηλεκτρονικής επίδοσης νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσω εδώ αλλά αυτό τέλο πάντων είναι μια γεύση των συζητήσεων που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα για την επίδοση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, ε, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μου. Είμαι Ζουλ Κιλιμπέρη από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, καθηγητής ε, και είμαι εισηγητής ε, για την ομάδα εργασίας ε, προσωρινά μέτρα και μέτρα προστασίας από το Πανεπιστήμιο Ζάμπρεν και με τέσσερις άλλες ομάδες εργασίας ε, που έχουν 6 με 8 μέλη που είναι είτε επαγγελματίες είτε ακαδημαϊκοί διότι θέλουμε να έχουμε και ανθρώπους από όλες τις κατευθύνσεις αλλά και από όλη την Ευρώπη. Δεν θα μπω στα γενικά σημεία που ήδη έθεσε η συνάδελφος Εύα. Θα επικεντρωθώ στο δικό μου θέμα, τα προσωρινά μέτρα και μέτρα προστασίας. Εμείς θέλουμε να καλύψουμε μια μεγάλη ποικιλία τέτοιων μέτρων, τα οποία θεωρούνται ε, ως πολύ σημαντικά σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή πάγωμα, κατάσχεση ή ε, προσωρινά μέτρα ε, για να γίνει ή να μην γίνει κάτι ε, σε διαδικασίες ας πούμε ψυχοφάντησης αν θέλεις να ανασταλεί μία δημοσίευση πριν κρυθεί η ουσία της υπόθεσης θεωρούμε ότι τα ασφαλιστικά μέτρα μπορεί να είναι για παράδειγμα η λύση επίσης διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων η αποκάλυψη πληροφοριών κάτι πολύ αποτελεσματικό που γίνεται πολύ στην Αγγλία και όχι τόσο στην υπόλοιπη ε, Ευρώπη και προσωρινές πληρωμές ενδεχομένως. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε κανόνες ε, οι οποίοι θα ρυθμίζουν κάθε ένα από αυτά τα διαφορετικά είδη προσωρινών μέτρων. Υπάρχει μια μεθοδολογία στους Ευρωπαίους νομοθέτες που έχει αποδεδειγμένη αξία στο παρελθόν και σήμερα. Ε, γενικά στην Ευρώπη τα προσωρινά μέτρα πάντοτε αντιμετωπίζονταν με έναν γενικό τρόπο, ας πούμε στα ε, έγγραφα των Βρυξελών ήταν πολύ γενικές οι διατυπώσεις, ε, γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένα λόγια και να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση ας πούμε στον όσον αφορά τη διατήρηση λογαριασμών και άλλα τέτοια ζητήματα. Ο σκοπός είναι να προσφέρουμε μία συγκεκριμένη ομάδα μέτρων για κάθε διάσταση αυτής της λειτουργίας και ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε και διάφορες επιλογές έτσι ώστε τα δικαστήρια στην Ευρώπη να έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν τις διάφορες πρακτικές και να επιλέγουν τα μέτρα που θεωρούν ότι βελτιώνουν τη διαδικασία τους και ε, στην ουσία ανταποκρίνονται στις ανάγκες ε, που υπάρχουν ε, και, που, και τις οποίες επιλύουν τα προσωρινά μέτρα. Παρόλο που η εντολή Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού δεν είναι απαραίτητα στα πλαίσια αυτού του πεδίου είναι ε, το αγγλικό αντίστοιχο του παγώματος ε, των λογαριασμών και της απόφασης για τη δέσμευση δηλαδή ε, και δεν θα πρέπει οι ομάδες να μην μπορούν να διερευνήσουν νέους δρόμους. Εμεί θέλουμε να τους προσφέρουμε νέα εργαλεία, να προσφέρουμε νέα εργαλεία στα διάφορα ε, δικαστήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, ο συνολικός στόχος είναι σίγουρα διτός. Καταρχάς, ε, να προωθηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία προσωνόμετρων στην Ευρώπη ε, εμποτίζεται σε μεγάλο βαθμό, κυρίως επειδή υπάρχει θέμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης δεν υπάρχει κυκλοφορία μέσα στην Ευρώπη και θεωρείται ότι μέσα από τη σύνταξη αυτών των κανόνων θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη διότι θα υπάρχουν ευέλτιστες πρακτικές οι οποίες στη συνέχεια θα πείθουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια ότι εύκολα θα εφαρμόζονται και θα αναγνωρίζονται τα προσωρινά μέτρα στις υπόλοιπες χώρες. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προόδου και σε επίπεδο υφιστάμενης νομοθεσίας. Ευχαριστώ, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γι' αυτό. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής κύριε. και κύριοι, είμαι ο Φερνάντο Νασκόν, καθηγητής νομικής στη Μαδρίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να παρουσιάσω ένα μέρος ε, το έργο για το οποίο είμαι υπεύθυνο. Είμαι συν εισηγητή τη ομάδα εργασία για τα θέματα των τεκμηρίων. Ένα μεγάλο μέρο ε, των ιδεών αυτών έχουν ήδη παρουσιαστεί από του προλαλήσαντε ε, συναδέλφου. Δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά. Θέλω να παρουσιάσω κάποιου κανόνε που αντανακλούν τι βέλτιστε πρακτικέ, λαμβάνοντα υπόψη και το κεκτημένο ε, δίκαιο της Ευρώπης και συγκριτικές εμπειρίες. Θέλουμε να έχουμε μια κοινή αντίληψη ανάμεσα στα δικαστικά ε, συστήματα που είναι πολύ διαφορετικά στον τρόπο οργάνωσης τους και λειτουργίας τους επί καθημερινής βάσης, όπως έχει ήδη λεχθεί. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να ε, προωθήσουμε παρόμοια πρότυπα σε ό,τι αφορά τη δίκαια ε, διαδικασία και την αποτελεσματική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τεκμήρια. Ε, η ομάδα που ασχολήθηκε με τα τεκμήρια έχει το ε, το πιο πλατή πεδίο εφαρμογής γιατί δουλεύουμε σε διάφορες κατευθύνσεις. Ξεκινάμε με ένα, μια κοινή σειρά από ε, κοινού κανόνες, κανόνες αποκλεισμού, ο των τεκμηρίων, ε, δικαιώματα και καθήκοντα των δικηγόρων και των δικαστών, ε, οι οποίε θα μπορούσαν να ήταν οι βέλτιστε πρακτικέ σε αυτό το τομέα. Στη συνέχεια θα δούμε κάποιου πιο συγκεκριμένου τομεί. Πρώτον, ε, πρόσβαση στα τεκμήρια και τις πληροφορίες που είναι ένα πολύ επίμαχο θέμα και κρίσιμο θέμα διότι η κουλτούρα που επικρατεί είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Δεν έχουμε την ίδια αντίληψη για το πώς μπορεί να γίνει η πρόσβαση στα τεκμήρια, στα στοιχεία, στις αποδείξεις των ε, διαδίκων. Κάποιες ε, κουλτούρες είναι διαφορετικές όπου ε, επιδεικνύονται τα τεκμήρια ή δίνονται, επιδίδονται στοιχεία ή έγγραφα που δεν θα έπρεπε. Ο νόμος, ε, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ε, πάει προς άλλη κατεύθυνση ό,τι αφορά τα, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησία. Θα πρέπει να υπάρχει μια χρυσή τομή ανάμεσα στις, στα συστήματα και στα θέματα εμπιστευτικότητα βέβαια και θα δούμε επίσης και ε, το, την καρδιά των κανονισμών σχετικά με τα τεκμήρια που θα είναι ο καλύτερος τρόπος ε, ακρόασης των ε, μαρτύρων ή εξασφάλισης τα τεκμηριών και μαρτυρίας από εμπειρογνώμονες. Αυτά ήθελα να πω. Thank you, Mr. Chairman. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίε και κύριοι. Είμαι ένα Βενετσιάνο, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Ινστιτούτου Ενωπήσης του Ιδιωτικού Δικαίου, UNIDROIT. Ε, συμμετείχα μαζί με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, Δικαίου. Ε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς ε, τον Πρόεδρο και την Επιτροπή που μας δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτό το κοινό έργο. Πιστεύουμε ότι ε, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό έργο από πρακτική άποψη, διότι επηρεάζει την επαγγελματική και την προσωπική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ήλαϊτ που ανέλαβε την πρωτοβουλία να βρεθούμε εδώ. Το UNIDROIT είναι ένας Παγκόσμιος Οργανισμός ε, αποτελείται από 63 κράτη-μέλη, τα περισσότερα είναι ευρωπαϊκά, έχουμε ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία στους κόλπους του UNIDROA. Παρά ε, το παγκόσμιο χαρακτήρα, η UNIDROA ήταν πάντα ανοιχτή στην ιδέα της περιφερειακής εναρμόνισης, όπως ε, εκφράζεται ρητός στο καταστατικό μας έγγραφο. Και γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό το project, αυτό το έργο. Για μας αυτό το project έχει δύο στόχους. Πρώτον είναι να επιδιώξουμε μια συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας. Και δεύτερον ε, η ιδέα ε, που ξεκίνησε από τις αρχές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου και της UNITRO που ε, από την αρχή ε, έπρεπε να συμπληρώνονται από περιφερειακούς κανόνες και είναι για μας ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και η ιδέα είναι να δούμε κατά πόσο και σε ποιο βαθμό αυτές οι αρχές είναι συμβατές με τις ε, ευρωπαϊκές νομικές παραδόσεις, πιστεύουμε ότι είναι, αλλά και πώς θα μπορούσαν να συμφέρουν έτσι ώστε να πετύχουν ένα πιο συνεχτικό σώμα κανόνων, χωρίς να διαγράψουμε βέβαια τις εθνικές ιδιαιτερότητες, αν θεωρούνται ε, να είναι σημαντικές. Ε, εν συντομία και κλείνοντας, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να έχουμε ένα ε, εργαλείο soft law για τους θεσμούς, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό αυτή η ακρόαση είναι πολύ σημαντική για, για μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα πέντε μέλη, τους φιλοξενούμενους μας, για τις παρουσιάσεις τους και αν ε, μας επιτρέπετε μπορεί να υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις προς εσάς. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Εγώ έχω μια ερώτηση. Υπάρχει κάποιο χρονικό χρονοδιάγραμμα αυτού του προγράμματος, πότε ε, να αναμένουμε τα αποτελέσματα κλπ. Πρώτα απ' όλα ακούσατε τις τρεις αρχικές ομάδες εργασίας. Έχουμε άλλες δύο που ξεκίνησαν να δουλεύουν παράλληλα. Ελπίζουμε να έχουμε κάποιο σχέδιο κανόνων από αυτές τις τρεις ομάδες στις αρχές του ερχόμενου χρόνου αλλά το όλο πρόγραμμα έχει προθεσμία να λήξει μαζί με το πρόγραμμα της UNITROA το 2017. Αλλά θα είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία και θα, μας, θα είναι χαρά μας να σας δίνουμε αναφορά ε, στην διαδικασία αυτή για την πρόοδό μας. Αν θέλετε να παρακολουθείτε την πρόοδο, βέβαια, φυσικά λέει ο Πρόεδρος από τη συνάδελφη, από τα μέλη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Δεν ε, βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Σημαίνει ότι η παρουσιάση σας ήταν ε, ε πλήρης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που παρουσιαστήκατε εδώ και μας συγχωρείτε πάρα πολύ για την καθυστέρηση που προκλήθηκε με την αλλαγή στην μερίσια διάταξή μας. Ήταν μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και προσβλέπουμε ε, στην ε, παρακολούθηση της πρόοδου του έργου σας. Σας ευχαριστώ πολύ. This was point number 13 and... Αυτό ήταν το σημείο υπερθμό 13, περνάμε τώρα στο υπερθμό 14. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. σχετικά με προστασία της αναγνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται εμπορικών απορρίτων. Πιστεύω πως ε, το λόγο θα πάρει η συγγήτρια κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα έχουμε την τέταρτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πάνω στο ζήτημα της προστασίας τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών προφορών που δεν αποκαλύπτονται και με την σημερινή ανταλλαγή απόψεων θα ξεκινήσει επισήμως ε, η διαδικασία για να χαράξουμε τον δρόμο που θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε στην έγκριση της εκθέσεώς μας σε αυτό το σχέδιο οδηγίες. Έχουμε λοιπόν αυτήν την, αυτό το εγχείρημα το οποίο και οι μεν και η δε που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση και οι σκιώδεις συζητήτες φυσικά θα μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε τις θέσεις μας και μια ακόμα φορά ως συγγήτρια της Επιτροπής Δομικών Υποθέσεων θα μπορέσω να προχωρήσω στην εξέταση των τροπολογιών, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να τις ε, ψηφίσουμε στις προσεχείς ημέρες. Σας είπα ότι η έκθεσή μου, όπως ε, την έχετε λάβει, επιθυμεί να είναι ισορροπημένη. Ευαίσθητη ισορροπία, το αντιλαμβάνομαι, αφενός ε, από την προσφορά μιας προστασίας, μιας ασφάλειας αποτελεσματικής για τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό, ο οποίος συχνά είναι παράνομος μέσω μιας πανοπλίας μέσων και μέτρων ουσιαστικών. Και αφετέρου γνωρίζουμε πως ε, υπάρχει ανάγκη διατήρησης σημαντικών θεμελιωδών ελευθεριών. Σκοπός ε, της εργασίας μας ε, βρίσκεται στην ευθεία γραμμή που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο χρήσιμο για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας προστατεύοντας αυτό το άειλο προνόμιο που συχνά είναι η καινοτομία, η έρευνα και ούτω καθεξής. Οι τροπολογίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν καταληφθεί μέχρι τις 18 ε, ε, Μαρτίου κάτι το οποίο μας επέτρεψε να τις λάβουμε υπόψη μας και να μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες. Είναι 302 οι τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν. Από εσά αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ήθελα σε αυτό το στάδιο να καταθέσω νέες τροπολογίες, δηλαδή να τροποποιήσω το σχέδιο έκθεσής μου. Δεν το θεώρησα απαραίτητο εν ώψη των ε, ανταλλαγών απόψεων που έχουμε ήδη κάνει και να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων για τις ε, προτάσεις τους και τις τροπολογίες τους, ε, οι οποίες ε, είναι ουσιαστική σημασία και αυτό θα το δούμε στο πλαίσιο των συζητήσεων, των μελλοντικών συζητήσεων. Χαίρομαι που σχεδόν το σύνολο των τροπολογιών που κατέθεσαν δεν θέτουν αμφιβόλου την αρχή της καταλληλότητας της νομοθεσίας, την αρχή και της καταλληλότητας ενός κειμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ούτε απαρνούνται τον, ε, τους μηχανισμούς. Αυτό μου επιτρέπει να εργαστώ ε, με όρους ευνοϊκούς ε, και να ξεκινήσω μια διαπραγμάτευση η οποία θα έχει αίσιο πέρασε. Να κάνω λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις ε, επί ουσιαστικών σημείων που εγώ ίδια πρότεινα και καταρχάς να κάνω κάποια αρχικά σχόλια των βασικών τάσεων όπως ε, τις είδα εν ώψη της πρώτης ανάγνωσης ε, και σύμφωνα με τις 300 κέντρο πολίτου κατρυφή. Τώρα να υπενθυμίσω πράγματα που είχα ήδη την ευκαιρία να πω, τα επαναλαμβάνω λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό η προστασία του, του σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εξωθεί με την δημιουργία ενός δικαιώματος πνευματικής διοκτησίας. Δεν είναι κάτι που θέλησε να προτείνει η Ευρωπαϊκή Ευρωπή και είμαι απολύτως σύμφωνη. Δεν πρόκειται λοιπόν για τη δημιουργία ενός νέου δικαίου πνευματικής διοκτησίας. Αυτό διατρέξει όλες, όλες, το, όλες τις εργασίες μας. Κάποιες επιστροπολογίες που έχουν κατατεθεί αμφισβητούν μια κάποια σημειολογία, κάποιες, κάποια ορολογία με την έννοια ότι αφορά στον τομέα της πνευματικής διοκτησίας κρίνω, αλλά αναφίβολα θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε, πως τίποτα δεν μπορεί να Ε, θεωρηθεί ότι αυτή η ορολογία περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτόν τον τομέα της σημαντικής διοκτησίας. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε διότι υπάρχουν τροπολογίες ε, που αφορούν το θέμα. Μια άλλη σημαντική τάση που διαπίστωσα στο πλαίσιο αυτής της πρώτης ανάλυσης των τροπολογιών αφορά τη συμπερίληψη και την στήριξη του δημοσίου συμφέροντος απέναντι στις ε, εμπορικές, στα εμπορικά απόρριτα. Να πω ότι το σχέδιο της έκθεσής μου τονίζει τις ανάγκες ε, της διαφάνειας που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και που προκύπτουν από το ενωσιακό δίκαιο ή από τα εθνικά δίκαια υποχρεώσεις διαφάνειας όπου ουδής ε, μπορεί να ε, παραιτηθεί και αυτό είναι σαφές και στο κείμενό μου αναφέρεται ρητά. Ουδής λοιπόν μπορεί να παραιτηθεί στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας ε, για την ε, επαγγελματική τεχνογνωσία. Αναφέρεται αυτό αναφέρεται στα άρθρα στα τροπολογίες 100 και 24. Το γενικό συμφέρον θα πρέπει να υπηρεσχεί στο πλαίσιο των εμπορικών, από το εμπορικό απορρίτου, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει που αποτελεί και την δημοκρατική έκφραση. Είναι σαφές λοιπόν πως τίποτα δεν θα πρέπει να μπορεί να παρακάμψει αυτή την αρχή. Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε. Ξέρω ότι αυτό θα χρειαστεί χρόνο, αλλά πρέπει από των ζητημάτων αυτών, δημόσιο συμφέρον, ε, γενικό συμφέρον, να βρούμε συμβαστικέ λύσεις. Να επαναλάβω ότι αυτό το σχέδιο οδηγία ήθελα να να γίνει σαφές που σε περίπτωση που είναι δεκτή η οδηγία να θα υπάρξουν ε, κάποιες αλλαγές στα κράτη-μέλη δεν θα μπορούσε να γίνει καμία παράκαμψη ουδενός μέτρου ειδικά των εξαιρέσεων ε, που προβλέπονται στην λόγω οδηγία, εάν και εφόσον εγκριθεί, από τα κράτη-μέλη, όταν θα βρίσκονται στη διαδικασία της ε, μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Αυτό αποτελεί μια νομική ασφάλεια την οποία ήθελα να συμπεριλάβω. Τώρα φτάνω στο άρθρο 4. Άρθρο 4 παραγωγός 2 που είχε ως αποτέλεσμα να κατελευθούν πολλές τροπολογίες. Εστιάζει λοιπόν άρθρο 4 παράγραφος 1, παράφη 1 και 2 και ειδικά στην παράγραφο 2 δεδομένου ότι πρόκειται για τις παρεκκλήσεις Έγιναν λοιπόν πολλές συζητήσεις και προέκυψαν πολλά ερωτήματα. Αφορούν την ελευθερία της έκβασης και την ελευθερία της πληροφόρησης. Το επαναλαμβάνω λοιπόν ρητά πως ο στόχος είναι να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο πληροφόρησης και υψηλό επίπεδο κυκλοφορίας των πληροφοριών στην κοινωνία μας και στην οικονομία μας. Νομίζω πως είναι προφανές, ίσως χρειάζεται να το τονίσουμε, βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, είναι η οικονομία της γνώσης που βρίσκεται στην βάση της αργοριστικότητας της οικονομίας μας και δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένας περιορισμός στην κυκλοφορία των προφοριών, της γνώσης και το επαναλαμβάνω επίσης σε μια δημοκρατική κοινωνία θεμελιώδεις ελευθερίες αποτελούν την πολύτιμους λήθους που θα πρέπει να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε στις τροπολογίες 6-8 υπενθυμίζω μία σειρά από που αφορούν αυτέ τι θεμελιώδει ελευθερίες που είναι ελευθερία της έκφρασης, ελευθερία της πληροφόρηση, τροπολογίε 6 και 7 λοιπόν. που κάποιοι θεμητά μπορούν να κρίνουν ότι μπορούν να τύχουν περαιτέρω βελτίωσης. Αναφέρονται λοιπόν στις τροπολογίες ελευθερία πληροφόρηση, τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, προστασία του μυστικού, των, του απόρριτου των πηγών. Αναφορές λοιπόν στα θεμελιώδη δικαιώματα διατυπώνονται ρητά. Αυτά τα θέματα λοιπόν, αυτοί οι λόγοι προκάλεσαν ε, πολλές τροπολογίες, τις οποίες θα εξετάσω με προσοχή και φυσικά θα κοιτάξουμε από κοινού αυτές τις τροπολογίες ε, διότι θεωρώ ότι με καλή θέληση και με την κατάλληλη εργασία έχουμε τους τρόπους ε, να βρούμε δίνοντας επικοδομητικό πνεύμα η μεν και η δε να βρούμε λοιπόν τις καλές διατυπώσεις και τους καλούς συμβασμούς τόσο πάνω στο ζήτημα αυτό όσο και πάνω σε άλλα. Αν και αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, άρα πιο ευαίσθητο και δύσκολο να το μεταχειριστούμε, να το αντιμετωπίσουμε. Προσεγγίζω λοιπόν στο τέλος ε, το παρέμβαση του πρόεδρο. Πρόεδρε, αναφέρομαι σε μια... ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει στο παρελθόν πολλές ε, που προσπάθησα να επικαθέσω τροπολογίες, πρόκειται για το ζήτημα της κινητικότητας των εργαζομένων και των φόβων που εκφράστηκαν για ενδεχόμενα φραγμούς στην ελευθερία κυκλοφορίας των εργατών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για τις προσπάθειές τους και να πω πως ε, η λόγω οδηγία παρουσιάζει κάποιες ε, τροχοπέδες, θα έλεγα, κάποιους φραγμούς, κάποια αποτρεπτικά μέτρα για τους ε, εργαζόμενους ε, με υψηλή δίκευση. Έλαβα υπόψη μου τους φόβους που εκφράστηκαν και πάνω στο θέμα αυτό θα είμαι ευτυχής να το εμβαθύνουμε και να συζητήσουμε τους ηγητές των ε, πολιτικών ομάδων έτσι ώστε να κάνουμε μια χρήσιμη αξιολόγηση και βελτίωση του κείμενου της οδηγίας και κλείνω με το συγκεκριμένο ερώτημα του προθεσμίας διαγραφής ή ε, παραγραφής Αυτά, τα, αυτά που τα οποία προέκυψαν από τις ε, αποφάσεις που έλαβαν οι δύο επιτροπές ε, προστασία κανολωτών και ε, βιομηχανίες και έρευνες μεταξύ των τροπολογιών που έχουν καταθέσει το δύο αυτές τροπολογίες οι επιτροπές συγγνώμη, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες τώρα στο σχέδιο εκθέσεώς μου γνωρίζετε ότι ήθελα να υπάρξει σαφής απόφαση περί του δικαιώματος παραγραφής ε, με ένα όριο τριετίας. Αυτό προτείνω στην τροπολογία με περίπτωση 28. Άλλες ε, επιλογές υπάρχουν ακόμα επιτάπητος. Εγώ ήθελα κάτι το απλό, το εύπεπτο που προκαλεί την ε, εναρμόνιση. Ξέρετε ότι στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να υπάρξει εναρμόνιση σε τι αφορά την ε, επαγγελματική γνώση. Ήθελα λοιπόν να προκύψει αυτή η ε, εναρμόνιση αυτή τριετής προθεσμία που προτείνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΜΚΟ και εδώ ευχαρίζω να το συζητήσω με τους συναδέλφους αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε σε κάποιο σημείο τον Κέρσορα. Και μια ακόμα πρέπει να ε, υπάρχουν διασφάλιση διασφαλίσεις και να δώσουμε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπλα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ε, με τα ίδια όπλα εταιρείε ε, που είναι πραγματικά κυνηγοί, είναι θύτες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε όλες τις ε, προϋποθέσεις διατήρησης των μηχανισμών αλλά και να μπορέσουν αυτοί οι μηχανισμοί να είναι λειτουργικοί, αποτελεσματικοί και να τεθούν σε ισχύ και εφαρμογή. Αυτά λοιπόν, ελπίζω τις προσεχείς εβδομάδες ε, να έχουμε ικανοποιητικές και επικοδομητικές συζητήσεις ε, για να καταλήξουμε μια συμφωνία όσο πιο στεναρή γίνεται. Κρατώντα όμω την κατεύθυνση που ανέφερα, δηλαδή προστασία της καινοτομίας και της ε, προστασία της αεραγωνιστικότητας των, Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκής Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πολύ περιεκτική παρουσίασή της. Έχουμε καταθέσει αρκετές τροπολογίες και η πρόταση έχει ακόμη δρόμο να διανύσει μέχρι να γίνει αποδεκτή. Ορισμένα από τα προβλήματα που είναι αρκετά σημαντικά για μας έχουν ήδη εγερθεί στις επιτροπές γνωμοδότησης που έχουν εμπλακεί και θα ήθελα να τα τονίσω. Πρώτον, είναι το θέμα του πεδίου εφαρμογής του τι μπορεί να αποτελεί εμπορικό μυστικό. Αυτό είναι πολύ πλατή. Ε, δεν είναι αναγκαίο να δούμε τον ορισμό απλά από τη Συμφωνία TRIPS, διότι αυτός ο ορισμός έγινε σκόπιμα για να περιλάβει ε, μια, ένα μεγάλο φάσμα παραδόσεων και τρόπων προστασίας του εμπορικού μυστικού στα προσυπογράφοντα κράτη. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός προστασίας των πληροφοριών ε, αν υπάρχει νόμιμο εμπορικό συμφέρον προστασίας αυτών των πληροφοριών. Πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ψευδών ε, ισχυρισμών, απαιτήσεων. Κάποιες μεγάλες εταιρείε μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την προστασία εμπορικού μυστικού για να ε, κρατήσουν έξω αθέμητο ανταγωνισμό. Και ε, το θα πρέπει να μπορεί να, να αποδεικνύεται ότι έχει λάβει χώρα πραγματικά μια παρανομή αποκάλυψη εμπορικών μυστικών και ε, κάποια προληπτικά μέτρα που ήδη δημιουργούν ε, στοιχεία προτού ένας ε, δικαστής αποφανθεί ότι έχει πέρθει αποκάλυψη μυστικών. Σχετικά με το άρθρο 4, δεν βλέπουμε γιατί από τη μια πλευρά στο πρώτο μέρος μιλάμε για την νόμιμη απόκτηση ε, ε, ε, είναι νόμιμη, αλλά για τη χρήση και αποκάλυψη για την ελευθερία της πληροφορήσης δεν υπάρχουν ένδικα μέσα. Όταν εφαρμόζεται κάποια εξαίρεση θα, θεωρεί, θα πρέπει να θεωρείται και αυτή μια νόμιμη αποκάλυψη. Για την περίοδο περιορισμού πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η κινητικότητα των εργαζομένων έτσι ώστε αυτή η περίοδος να είναι βραχία ιδιαίτερα για εργαζόμενους, πρώην εργαζόμενους, δεν πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος, διότι αλλιώς δεν θα είναι δυνατόν αυτοί πραγματικά να έχουν την ασφάλεια δικαίου όταν μετακινούνται από μια εταιρεία σε άλλη. Κάτι άλλο το οποίο είμαστε σε καλή οδό, αλλά μπορούμε να το διευκρινίσουμε, είναι ότι πράγματι δεν μιλάμε για διανοητική ιδιοκτησία. Οι πραγματικές διαφορές ε, για παράδειγμα, αν υπάρχει δίπλωμα ευρασιτεχνίας, το δικαίωμα είναι χαρακτηριστικό της ίδιας τη πληροφορίας. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι το εμπορικό μυστικό έχει προστασία μόνο και μόνο γιατί ε, ε καθ' την περίοδο που είναι μυστική αυτή η πληροφορία. Και αν υπάρχει ανεξάρτητη ανακάλυψη αυτών των πληροφοριών. Όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί στις διαπραγματεύσεις της TTIP ε, συζητώνται ε, μυστικά στο θέμα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει σαφές ότι η νόμιμη αποκάλυψη των, των μυστικών περιλαμβάνει πληροφορίες που απαιτούνται δια ή από κάποια επίσημη αρχή ότι δεν είναι κάτι όπου μια κυβέρνηση θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι απαντώντας ε, σε ένα αίτημα ελευθερίας ε, πληροφόρησης θα μπορούσε να αποτελέσει παράνομη αποκάλυψη εμπορικών μυστικών. Θα πρέπει αυτό να καταστεί σαφές. Επίσης, προστασία των εργαζομένων και διασφάλιση ότι δεν υπάρχει ε, αλόγιστο άχθος στους εργαζομένους και επίση θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν ε, περιττό ε, φόρτο εργασίας. Για το θέμα της προστασίας των καταγγελτών πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταστεί ότι η παράνομη αποκάλυψη ενός εμπορικού μυστικού θα πρέπει να περιλαμβάνει ε, μια πρόθεση οικονομικής πρόκλησης ζημιάς Εάν αποκαλύπτονται μυστικά για το δημόσιο συμφέρον, αυτή δεν είναι παράνομη αποκόλληψη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ε, μιλάμε για θέματα πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος, για παράδειγμα για ε, ζημιά στο περιβάλλον, όπου αυτός που κρατάει το μυστικό μπορεί να μην παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει σημαντικό δημόσιο συμφέρον. Σημαίνει ότι ο θα ε, πρέπει να είναι σε θέση να δίνει αυτές τις πληροφορίες στον τύπο για παράδειγμα. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά, οι πιο σημαντικές προτεραιότητες στις διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε ότι στην διαδικασία συμβιβασμού θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια κοινή θέση. Ευχαριστώ. Ε. Σας ευχαριστώ εγώ. Η κυρία Γκούτλαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Λαγκρίπ και για τη σκληρή δουλειά και για αυτή την μακρά ε, παρουσίαση του θέματος. Είναι σημαντικό νομοθέτημα αυτό, γι' αυτό είναι κρίσιμο να το πετύχουμε σωστά. Γι' αυτό βλέπετε και μια τέτοια μεγάλη σειρά τροπολογιών. Γιατί θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό νόμο. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι χάρηκα που άκουσα ότι είναι ε, σημαντικό να ληφθεί υπόψη η κινητικότητα των εργαζομένων. Ε, θα ήταν καλό να βρεθεί μια λύση εδώ, διότι είναι σημαντικό να μην μειώσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Ε, πρέπει να γίνει κάτι σε αυτό το τομέα και πραγματικά χαίρομαι που το αναφέρατε και ελπίζω να βρεθεί μια χρυσή τομή εδώ. Επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι στηρίζουμε την διαφάνεια ε, για θέματα έρευνας και περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, συλλογή στοιχείων σε θέματα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δεν πρέπει αυτή η πρόταση να παρεμποδίσει τις έρευνες ε, ούτε στο τομέα της ιατρικής αλλά ούτε και στη διαδικασία μιας αηφόρου κοινωνίας. Για ε, σκοπούς ασφάλειας είναι σημαντικό αυτό που είπε και η κυρία Ριέντα σχετικά με ε, τους καταγγέλτες. Δεν μπορεί να τιμωρείται κανείς στα πλαίσια αυτής της ε, οδηγίας. Θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να μεταδίδονται στα μέσα ή στις ε, αρμόδιες αρχές κάποια, κάποιες πληροφορίες. Στηρίζω τις τροπολογίες που λένε ότι θα πρέπει να ε, πρόκειται για οικονομική ζημιά προς μια εταιρεία γιατί όταν γίνεται για θέματα ασφάλειας ή για την πρόληψη του εγκλήματος είναι σημαντικό να μην αισθάνονται το φόβο να το καταγγείλουν. Επίσης θα ήθελα να δω μια καλύτερη διατύπωση των συλλογικών συμβάσεων και έχουμε κάποιες τροπολογίες στο θέμα αυτό και αυτό είναι το δικαίωμα των συνδικαλιστών και εκπροσώπων και τη δυνατότητα των εθνικών δικαστηριών να ρυθμίσουν οποιασδήποτε αποζημιώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την νομική πρακτική. Είναι κάποια λοιπόν από τα θέματα σχετικά με τις δικές μου τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιθυμώ να ευχαριστήσω ειλικρινά την εισηγήτρια για την εργασία της αλλά και για την ε, διαθεσιμότητά της, την, προθεσμία, την προθυμία της που ανέφερε και προ λίγου προκειμένου να συνεργαστούμε για να αποκτήσει ένα ψηλό προφίλ αυτή η οδηγία. Γνωρίζουμε πως υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από το ζήτημα, ζήτημα το οποίο πρέπει να είναι σαφές ε, για να αποφύγουμε μελλοντικές ε, παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Ε, σε ό,τι αφορά την ομάδα μου, σα σας επιβεβαιώνω τις αρχές που προκύπτουν από τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα που αφορά στην στο know-how, την τεχνογνωσία και του εργαζόμενου. Και δεν μιλάμε μόνο για την κινητικότητα που είναι πολύ σημαντική για τι επιχείρησει, αλλά μέσω των γνώσεων τα πρόσωπα αποκτούν μια συμβατική ε, ισχύ που του επιτρέπει να επιλέξουν άμεσα στι διάφορε εργασίε που του προτείνονται, αλλά και να ε, προσδιορίσουν τη σχέση τους και τις προϋποθέσεις της εργασίας. Είναι φυσικό ότι αν δεν υπάρχει σαφής εγγύηση και αν προσπαθούμε να τραγουδήσουμε την γνώση σε μυστικό, σε απόλυτο, τότε θα επηρεαστεί τόσο η κινητικότητα αλλά και η αξιοπρέπεια των προσώπων για την εργασία την οποία καλούνται να αναλάβουν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά που είπατε σήμερα είναι πολύ σημαντικά, θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται, αλλά γι' αυτό χρειάζεται μια αναφορά συνεπής σε ό,τι αφορά τις αρχές. Επίσης είναι σημαντικό να ε, θεσπίσουμε το γεγονός ότι το γενικό συμφέρον είναι υπεράνω και εκτός και πέραν του απορρίτου, ξεκινώντας από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και τις δημόσιες, διότι αν δεν ανταποκρίνονται ε, στους ε, ενδιαφερόμενους και τότε ο κίνδυνος ε, του να υπάρξουν μορφές ε, ανταγωνισμού παράνομες ε, είναι σημαντικός αυτός ο κίνδυνος. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε την διάκριση και να μην υπάρχει μια θεά περιοχή, θεά ζώνη. Έως εκ τούτου είναι απαραίτητο να γίνουν γνωστά αυτά τα στοιχεία που αφορούν σε Τώρα η ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης, προφόρησης, όπου αναφερθήκατε, ρυθμίζεται και από άλλα νομοθετήματα της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν μια δουλειά σχετικά απλή, διότι οι μνήες ε, είναι ήδη γνωστές όπως και ο ορισμός ε, του εμπορικού απορρίτου, σύμφωνα με τα όσα είπαν και κάποιοι συνάδελφοι, μπορεί να προσδιοριστεί και να οριστεί εύκολα και άρα με θετικές επιπτώσεις. Δεν θα πρέπει να κάνουμε αναφορά στον γενικό χαρακτήρα που μας οδήγησε μέχρι εδώ, αλλά να καταβάλουμε προσπάθεια για να έχουμε μια πιο σαφή ε, ε, πιο σαφή ορισμό του ζητήματος και να πω επίσης ότι αυτό το λεπτό σημείο των χρόνων παραγραφής και αναφέρομαι λέγοντας ότι έχω συμμετάσχει στην συνεδρίαση της ΣΥΜΚΟ ως ε, σκιώδης ηγητής. Εσείς προτείνετε τρία έτη. Κάποιοι έχουν προτείνει εξαετία. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Για δύο λόγους. Δηλαδή να αποφύγουμε ότι αυτό ε, θα αποτελέσει εμπόδιο στην κινητικότητα όπως αυτό που άπτεται με το ζήτημα της τεχνογνωσίας είναι ότι υπάρχει μια διαφωνία στο εξή ότι όσο μακρύτερο είναι η χρονική περίοδο τότε πιο δύσκολα είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος διότι αλλάζουν οι παράμετροι στην αγορά. Εάν λοιπόν έχουμε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα παραγραφής, έχουμε ένα παραπάνω πρόβλημα από την πλευρά της επιχείρησης. Δεν μπορώ να το αποκρίσω αυτό, αλλά μια αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη για τον χρήστη στην περίπτωση αυτή που είναι ο εργαζόμενος. Γι' αυτό λοιπόν τονίσαμε και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Φυσικά η λύση ήταν άλλη φύση. εξάλλου η πλειοψηφία στην Δημοκρατία έχει πάντα δίκιο. Ζητώ λοιπόν να υπάρξει μια περαιτέρω, ένας περαιτέρω προβληματισμός για το ζήτημα αυτό της παραγραφής, διότι ο περιορισμός ε, της παραγραφής, της διάρκειας παραγραφής θα έχει ε, θετικά αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα που πρέπει να προστατεύονται και να γίνονται σεβαστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ροζιέρ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Να χαιρετήσω την εργασία της εισηγήτριας ε, και το πνεύμα μέσα ε, στο οποίο ε, γίνεται αυτή η συζήτηση. Ο Σέρτζο Κομφεράτη συνόψισε τις μεγάλες γραμμές της ομάδας μου και εγώ ίδια έχω καταθέσει κάποιες τραπολογίες για να προστατεύσουμε την τεχνογνωσία των επιχειρήσεων αλλά και να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι ενώ έχουμε μια επικαιρότητα η οποία έχει φέρει πάρα πολλά θέματα στην, στο προσκήνιο αυτού του είδους ε, η, η λειτουργία είναι αυτή η λειτουργία που απαιτεί η δημοκρατία και ως εκ τούτου η θέση που θα πάρουμε πάνω στο θέμα μας οδηγεί στο να πούμε ότι η ελευθερία έκφρασης, η ανεξαρτησία, η ενημέρωση είναι στοιχεία της δημοκρατίας και της λειτουργίας αυτής και επιβεβαιώνουμε την αρχή ότι το δημόσιο συμφέρον ε, υπερισχύει Για το λόγο λοιπόν αυτό κρατήσει κάποιες τροπολογίες, ε, κάποια αφορούν στον ορισμό και για το άρθρο 4 που όπως ε, ελέγχθη ήδη προκαλεί πολλές συζητήσεις, θα πρέπει να είμαστε σαφείς στην προστασία ε, των εργαζομένων όταν οι αποφάσεις της επιχείρησης τους αφορούν Αυτές λοιπόν είναι οι γραμμές ε, των τροπολογιών που έχω καταθέσει. Είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να βρούμε μια κοινή θέση που θα επιβεβαιώνει τις μεγάλες αρχές των ευρωπαϊκών δημοκρατιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριος Μπεζεβέ από την Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Κομισιόν θα ήθελα να ευχαριστήσει την εισηγήτρια και τα μέλη για την επικοδομητική συζήτηση και τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Θα ήθελα να γύρω κάποια ζητήματα που ελπίζω να βοηθήσουν ε, τα μέλη στο να ε, επιτύχουν μια επικοδομητική συνένεση από αυτού. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε και η κυρία Ρέντα αναφέρθηκε ότι όλα τα κράτη-μέλη ήδη με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε αναλάβει δράση είναι ότι έχουν ασχοληθεί με διαφορετικούς τρόπους. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό το κείμενο που είναι βασισμένο στην εσωτερική αγωγή ε, ε, στην εσωτερική αγορά, με συγχωρείτε, και θα ήθελα ότι στις τροπολογίες δεν με εκπλήττει ότι βλέπω ότι υπάρχουν τροπολογίες για την ελάχιστη εναρμόνιση εκ μέρους της Κομισιόν θα έλεγα το ίδιο και στα κάτι μελη θα έλεγα το ίδιο όταν, μιλάς, όταν ζητάς για ελάχιστη ε, εναρμόνιση ε, πως κάτι σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Παρόλο που χρειάζεται, αυτό που πιστεύουμε έντονα είναι ότι αυτή η ρήτρα ελάχιστη εναρμόνιση δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των ασφαλιστικών δικλείδων που έχουμε θέσει μέσα στο κείμενο το να έχει μεγαλύτερη προστασία ε, εις βάρος των ασφαλιστικών ε, δικλείδων θα είναι αντιπαραγωγικό ε, στην ισορροπία που αναφερθήκατε όλοι, που είναι αναγκαία. Δεύτερον, αυτό το θέμα της ισορροπίας. Συμφωνώ με την εισηγήτρια και με τους άλλους ομιλητές είναι θεμελιώδες. Από τη μια πλευρά προσπαθούμε να διασφαλίσουμε, ότι, ε, να διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντα των ευρωπαϊκών χωρών στην διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους, ε, της δυνατότητας καινοτομίας και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, πλευρά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ε, τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα των εργαζομένων, των πολιτών και καταναλωτών είναι, ε, τυχάνουν πλήρους ε, προστασίας. Χωρίς να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, θα ήθελα να γύρω κάποια σημεία που ελπίζω να βοηθήσουν στο να πετύχετε μια ομοφωνή γνώμη. Πιστεύω ότι πολλά θέματα που έχουν γερθεί είναι θέματα που πιστεύουμε ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής αυτής της πρότασης. Για παράδειγμα, δεν πιστεύουμε ότι αυτό το κείμενο παρεμβαίνει, ούτε θα έπρεπε να παρεμβαίνει με τις εθνικές υποχρεώσεις που έχει η βιομηχανία να επικοινωνεί, να μοιράζεται ε, πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος στις δημόσιες αρχές. Δεύτερον, δεν πιστεύουμε ότι το κείμενο παρεμβαίνει καθόλου με τους κανόνες που υπάρχουν σχετικά με τη διαφάνεια συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των πολιτών να εξασφαλίσουν ε, κείμενα που είναι στην κατοχή των δημοσίων αρχών. Και τρίτον, δεν πιστεύουμε ότι το κείμενο και θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν πρέπει, να παρέμβαίνει με το, με το νομικό πλαίσιο των εργατικών σχέσεων και των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Το θέμα κλειδί που έχει γερθεί από τον κύριο Κουφεράτη, πιστεύω είναι ότι θέλουμε σίγουρα να εξασφαλίσουμε ότι η τεχνογνωσία και οι δεξιότητες των εργοδοτών δεν θεωρείται εμπορικό μυστικό. Έχουμε δει τροπολογίες που είναι ενδιαφέρουσες. Ε, θέλουν να προωθήσουν αυτό στο κείμενο. Είναι ουσιαστικό αυτό, πολύ σημαντικό σημείο. Υπάρχει ένα θέμα κλειδί. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρόταση ήταν σαφής, βέβαια πάντα χρήση βελτίωσης. Πιστεύουμε ότι ρήτρε αρνητικού πεδίου εφαρμογή θα πρέπει να ε, γίνουν και αυτό θα οδηγήσει το κείμενο να γίνει πιο απλό. Και αυτό θα είναι βασικό εάν το κείμενο αυτό θα μεταφερθεί σωστά στην ε, ε, χώρια νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό οι έννοιες του εμπορικού μυστικού ή του παραβάτη, της παράνομης ε, απόκτησης ή αποκάλυψης δεν πρέπει να ε, είναι ενάντια σε άλλες απαιτήσει ή να περιλαμβάνουν άλλες απαιτήσει που εμπίπτουν σε άλλους τομείς του δικαίου. Ένα άλλο σημείο. Δεν θέλουμε να δούμε αυτή την πρωτοβουλία να χρησιμοποιείται ε, ή να διαστρεβλώνεται για την ελεύθερη χρήση των πληροφοριών που είναι ε, δημοσιευμένες και που δεν θεωρούνται πια εμπορικά μυστικά. Είμαστε κατά νέων εξαιρέσεων στις βασικές ε, ελευθερίες. Άκουσα αρκετά σημεία σχετικά με το άρθρο 4 και τις εξαιρέσεις. Για να είμαστε απόλυτα σαφείς για το άρθρο 4 και ιδιαίτερα τις δύο διατάξεις 4, 1 και 2, 4.1. Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν περαιτέρω περιορισμού στα εμπορικά μυστικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να γίνει αυτή η διάκριση δηλαδή. Ε, σε σύγκριση με το 4.2, που είναι ε, μια παρέκκληση του, του άρθρου 3. Το κλειδί. Έχουμε μεγάλο σεβασμό ε, προς τους καταγγέλτες. Σήμερα οι καταγγέλτες και ε, ε, ε, αντιμετωπίζουν τον νόμο διότι ο καταγγέλτης είναι ο εργαζόμενος, δεν είναι ο δημοσιογράφος, είναι η πηγή. Αυτός που είναι μάρτυρας των πληροφοριών και που θα αντιμετωπίσει νομικές διαδικασίες διότι αυτός ή αυτοί το έχουν κάνει, το έχουν καταγγείλει κάποιες πληροφορίες. Αυτό το κείμενο, το τι κάνει, αναγνωρίζει το δικαίωμα του καταγγέλτη σε υπεράσπιση. Και είναι πολύ σαφές ότι κατά παρέκκληση, εάν πραγματικά διατηρεί το δημόσιο συμφέρον, τότε δρά ε, ε ένομα. Και στο 4-2 ε υπήρξε ανησυχία ότι είχαμε προτείνει συγκεκριμένα μια εξαρτή για το νόμιμο συμφέρον. Αυτό είναι ευρύτερο ακόμα από το δημόσιο συμφέρον. Περιλαμβάνει το δημόσιο συμφέρον και είμαι βέβαιος ότι τα μέλη, ελπίζω τουλάχιστον ότι όταν το εξηγήσω θα καταλάβετε ότι η αυτή η διασφάλιση είναι πάρα πολύ ε, δυνατή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το έργο που έχει πετελεστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το τέλος ε, της, του καταλόγου των ομιλητών. Η κυρία που θέλει να πει κάτι. Όχι. Πολύ σύντομα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, γιατί ήταν μεγάλη συζήτηση. Ευχαριστώ ε, τον καθένα σας. Ε, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να παραμείνουμε επικοδομητικοί και στο μέλλον να πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο για να μπορέσουμε να έχουμε όσο και το δυνατόν ευρύτερη συμφωνία γίνεται για να έχουμε μια συγκεκριμένη συνοχή και να ξέρουμε ακριβώς πού θέλουμε να φτάσουμε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε με αυτό το ανώτατο όριο να έχουμε μια κατεύθυνση και να μπορέσουμε να πορευτούμε ε, στο Στρασβούργο όπου θα γίνει μια πρώτη συζήτηση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προχωρούμε με έναν ικανοποιητικό ρυθμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Λεκρίτ. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος του σημείου 14 και συνεχίζουμε με το σημείο 15. Τώρα θα πρέπει να δώσω το λόγο στον εαυτό μου. Ε, θα σας δώσω τα στοιχεία σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένη συνένεση όσον αφορά στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής Διοκτησία και διοδράσης της ΕΕ που προτείνεται από την Επιτροπή. ω εισηγητή, αγαπητοί συνάδελφοι να πω το εξή. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έχουν καταθέσει τροπολογίες στο σχέδιο της έκθεσης Συνολικά ήταν 124 ε, τροπολογίες ε, και είμαι ευγνώμων διότι δίνουν μεγαλύτερη ακρίβεια στο κείμενο. Ε, πολλές φορές ε, στην ουσία θέτουν μια καλύτερη εικόνα, ε, δίνουν την ευρύτερη εικόνα και έχουν να κάνουν με τα ευρύτερα δημόσια συμφέροντα. Όπως ήδη ακούσατε θα υπάρχει μια συνάντηση των σκιωδών για αυτές τις ε, τροπολογίες και το σχέδιο έκθεση την επόμενη εβδομάδα την Τετάρτη. Ε, οπότε θα συζητήσουμε και τις ε, διάφορες τροπολογίες λεπτομερώς. Τώρα θα ήθελα να επικεντρωθώ στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής και να κάνω κάποιες προτάσεις για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας γενικότερα. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες, ειδικότερα αυτές που έχουν να κάνουν με την ιολογική σκέψη AD και τα άρθρα 6, 8 και 20. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι σε κάποιες γενικές δηλώσεις η κυρία Ντελβό έθεσε το θέμα την τελευταία φορά. Δεν ήθελα εγώ να δώσω κάποια νομιμοποίηση για κάποια παράνομη συμπεριφορά. Σε καμία περίπτωση δεν το ήθελα αυτό. Εγώ ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η, δυνα... η πραγματικότητα στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αν πρέπει δηλαδή να έχουμε μια ε, ε, εκστρατεία ευαισθητοποίησης των νέων για παράδειγμα. Θα ήθελα να συναντήσω τους ε, την επόμενη εβδομάδα. Αυτά. Από εμένα ζητώ, ε, και περιμένω τώρα να ακούσω ποιοι θέλουν να, ε, να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την εισαγωγή. Νομίζω ότι θα είναι δυνατόν να έχουμε αυτό το έγγραφο το οποίο έχει τόσο μεγάλο αριθμό ε, τροπολογιών. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το σχέδιο δράσης ε, για την επιβολή δικαιωμάτων ε, δια των ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να υπάρχει αποδοχή το λαό για το θέμα αυτό της διανοητικής ιδιοκτησίας ε, διότι ε, πρέπει στην ουσία να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σχετικά με την σημασία της διανοητικής ιδιοκτησίας να πω ότι υπάρχει ε, μια σχέση μεταξύ του ιδιωτικού δικαίου ε, αλλά και τη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων ε, και τον έλεγχο της ε, νομικής παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτή η ισορροπημένη σχέση είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη, της, υπόψη του το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα κλίμα ε, όπου υπάρχει περιορισμός ε, των ε, βασικών των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά ούτε και να ανοίγουμε τις πόρτες για την ποινικοποίηση των χρηστών. Για το δεύτερο θέμα υπάρχει παραβίαση των η εμπορική παραβίαση ας πούμε των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά υπάρχει και η ιδιωτική παραβίαση και η σχέση μεταξύ των δύο δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα διαχωρισμό, να δούμε ποια είναι τα θέματα ε, ε, παραβίασης από άτομα ή σε επαγγελματικό επίπεδο για να μην φτάσουμε σε ποινικοποίηση των χρηστών. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει ε, τήρηση των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν μιλάμε για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ε, και την ε, πνευματική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα του συγγραφέα, του δημιουργού μάλλον, είναι σημαντικό να έχουμε μια δίκαιη αμοιβή ας πούμε. Άλλο σημαντικό είναι η διερεύνηση η οποία θα βασίζεται σε τεκμήρια όσον αφορά στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Υπάρχουν τέτοιες έρευνες, όμως είναι κάπως ε, μεροληπτικές και θα πρέπει νομίζω να δούμε εμείς ως κοινοβουλευτικοί ε, κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια βάση για να μπορέσει ε, το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μέτρα για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ε, πρέπει να είναι ένα θέμα διαφανές, ε, να λάβει μέρος στο δημόσιο διάλογο όλος ο κόσμος και για μας αυτά είναι στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά και δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια κοινή θέση. Okay. Mr. Anderson. Άντερσον. Well, ήταν μια μεγάλη ημέρα και γι' αυτό θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Θα ήθελα να συνεργαστώ με τους άλλους Θεωρώ ότι χρειάζεται να υπάρχει κάποια ισορροπία για αυτό το θέμα. Ε, για τα θέματα που μπορούν να υπόκεινται σε δικαιώματα ευρεσιτεχνία ή όχι και μια ισορροπία σχετικά με τα διάφορα δικαιώματα που έχει ο καθένα. Υπάρχουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησία αλλά και ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της προσωπικής σφαίρας και θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του συστήματος του δικαστικού και θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην εμπλακούμε σε μια κατάσταση κατά την οποία αυτά τα δικαιώματα δεν ισορροπούν μεταξύ τους και πραγματικά ε, αδειμονώ να, να εργαστούμε σε αυτή την έκθεση. Ο κύριος Περσεβάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εκ μέρους της Επιτροπής για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα διάφορα μέλη που έχουν καταθέσει τροπολογίες. Ε, κάποια ε, σχόλια έχω τώρα σχετικά με τα όσα είπε και ο κύριος Κώστα για το την ανάγκη τεκμηρίων μέσα από το παρατηρητήριο και αυτό όχι υπάρχουν τώρα μελέτες οι οποίες γίνονται σχετικά με τα καλλιτικά που είναι αντικειμενικές δηλαδή με άλλα λόγια γίνονται ανεξάρτητα ε, και Υπάρχουν ε, συγκεκριμένα πλαστά προϊόντα στην αγορά, 10% εκτιμάται, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλα ε, στοιχεία και συνεργαζόμαστε με τον ΑΣΑ αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα στοιχεία και να επικεντρωθούμε στο θέμα το εμπορικό που έχει να κάνει με αυτήν την έκθεση κάτι ε, το οποίο αναφέρατε και με το οποίο συντασσόμαστε. Το δεύτερο στοιχείο που χαιρετίζουμε και είναι η ανάγκη που όλοι αναφέρατε να ληφθεί υπόψη οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναφέρατε και την ανάγκη καλής λειτουργίας του συστήματος δικαι... της δικαιοσύνης. Για την έκθεσή σας κύριε Πρόεδρε, να πω ότι δεν θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα του soft law απομονωμένα από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει και σε αυτό να ε, συμφωνήσουμε από άποψη τώρα διευκρίνησης. Εμείς στην Επιτροπή μας όταν μιλάμε για αυτόν τον νέο όρο, την προσέγγιση ακολούθησε το χρήμα, follow the money, δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με, το ε, με την προσέγγιση ακολουθήστε τον καταναλωτή ή τον πολίτη. Ε, στην ουσία εξετάζουμε ποιοι είναι οι εμπορικοί αυτοί, οι ποιες είναι αυτές οι εμπορικές οντότητες που βγάζουν λεφτά στην πλάτη των καταναλωτών. Και ε, να πω κάτι για τις τροπολογίες του κυρίου Κώστα. Δεν έχει να κάνει με τους ενδιάμεσους ε, που δρούν στο διαδίκτυο. Έχει να κάνει με όλους τους ε, ενδιάμεσους που έχουν να κάνουν με τις παραβιάσεις ε, σε εμπορικό επίπεδο. Θέλουμε να δούμε όλους αυτούς και να μπορούν ε, ε αυτοί που είναι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων να στραβούν κατά όλων αυτών των ενδιάμεσων. Τώρα για τη δίκαιη αμοιβή. Τα δικαιώματα σε δίκαιη αμοιβή. Όταν κοιτάμε την αρχή της αλυσίδας, εκεί λοιπόν που η, ε, ουσιαστικά οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ουσία παίρνουν κάποια αμοιβή, ε, βλέπουμε ότι αν ε, ε εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε περισσότερη προσφορά και αν δεν το αντιμετωπίσουμε σωστά μπορεί να μην υπάρχει αυτή η προσφορά λόγω έλλειψης κινήτρων. Προ... Προσβλέπουμε λοιπόν στις τροπολογίες σας και περιμένουμε την έκθεσή σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις. Εγώ προσωπικά πραγματικά δημονούσα για αυτή τη συζήτηση σχετικά με την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων και των αρχών που θα ε, περιληφθούν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα κλείσουμε τώρα λοιπόν με το σημείο 15. Είχαμε, έχουμε ήδη κάνει το σημείο 16. Οπότε να σας ενημερώσω ότι η επόμενη τακτική συνεδρίαση θα γίνει στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 6 Μαΐου και την Πέμπτη 7 Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στην Επιτροπή.